πρακτική που σαφέστατα αντιτίθεται στην στρατηγική τη Λισαβόνα για την παιδεία. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε να γίνεται κάτι τέτοιο σε κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Σα ευχαριστώ. Πραγματικά τελειώσαμε με αυτό το σημείο τη μεσή διάταξη. Σα ευχαριστώ για την κατανόησή σα, για την πειθαρχία που έπρεπε να επιδείξουμε και ελπίζω όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν, να μιλήσουν την επόμενη φορά. Οπότε τελειώσαμε με αυτό το σημείο. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, κοινή συζήτηση για δύο εκθέσεις. Σχέδιο προπολογισμού για το 2011 της κυρίας Σιντονιά Ελισβιέτα Γέντρεζιεύσκα, ελπίζω να μην έκανα λάθος το όνομά σας και μετά κατευθυντήριες γραμμές του προπολογισμού 2011 της κυρίας Τρίπελ για τα λοιπά τμήματα. Πρώτη λοιπόν έχει τον λόγο η κυρία Γετζεζεύσκα. Γιονσιγέσκα. Εν πάση περιπτώσει έχετε το λόγο για 8 λεπτά. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Komisarzu, Szanowne Koleżanki i Koledzy. Η διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2011 είναι ιδιαίτερα ιδιάζουσα, έκτακτη θα έλεγα, διότι είναι η πρώτη διαδικασία που θα εγκριθεί με τις αρχές της συνθήκης της Λισαβόνας. Είμαστε λοιπόν πιονέροι. Αυτό βέβαια έχει ναι, απαιτεί νέες υποχρεώσεις και από εμά. Και από εμά θα εξαρτηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διαθέτουμε αυτές, θα διαθέσουμε αυτές μας τις αρμοδιότητες. Εμείς θέλουμε να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας. Μία πρώτη καινοτομία είναι ότι δεν θα έχουμε δύο αναγνώσεις για τον προϋπολογισμό. Οπότε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν μία και μόνη ανάγνωση. Θα έχουμε λοιπόν μία πολύ σημαντική πρόταση, ε, πρόκληση μπροστά μας και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα πειθαρχημένοι διότι θα έχουμε μία και μόνη ευκαιρία. Δεν θα μπορούμε να έχουμε δεύτερη ανάγνωση. Οπότε εμείς στη συνδιαλλαγή θα πρέπει να εγκρίνουμε το μάξιμουμ κοινών σημείων. Η συνδιαλλαγή θα πρέπει να εκτιληθεί με πειθαρχία. Η Κομισιόν επίσης δεν κατάφερε να παρουσιάσει την ετήσια πολιτική τη στρατηγική γιατί διορίστηκε καθυστερημένα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρώτο θα εκφράσει τη γνώμη του, θα εκφράσει τα πρίμα λόγια για τον προϋπολογισμό του 2011 και αυτή είναι και η πρώτη σκέψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την έκθεση. Είμαστε οι πρώτοι λοιπόν που παίρνουμε το λόγο και όχι η Κομισιόν. Γιατί λοιπόν είναι ιδιαίτερο το οικονομικό έτος του 2011 στα πλαίσια του πολιετούς ε, ε, χρηματοδοτικού πλαισίου είμαστε στην πέμπτη χρονιά και μάθαμε ήδη πολλά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Στην Πολωνία λέμε ότι κουτουλήσαμε τον τοίχο, οι Άγγλοι έχουν φτάσει στο ταβάνι. Εμείς το εξαντλούμε αυτό το πολιετές πλαίσιο. Ε, τα περιθώρια είναι πραγματικά εξαντλημένα και οι δυνατότητες του Κοινοβουλίου να δράσει είναι ελάχιστες και περιορισμένες κυρίως ε, για το 1β, 1 εκατομμύριο και κάτι ευρώ και τη 2β 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχουμε πολλές δυνατότητες. Τώρα, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ζητά μια φιλόδοξη αναθεώρηση του ε, δημοσιονομικού πλαισίου, όχι γιατί μόνο τα περιθώρια περιορίζονται, αλλά γιατί η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις επιπτώσεις που θα έχει η συνθήκη της, ε, η της Λισαβόνας στο δημοσιονομικό πλαίσιο έχουμε νέες αρμοδιότητες ας πούμε για την ε, διαστημική πολιτική για την ε, εξωτερική πολιτική. Εμείς πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε το πώς θα υλοποιήσουμε την νέα στρατηγική του 2020. Αυτά τα σχέδια δεν τα είχαμε προβλέψει στο πολιετές μας σχέδιο. Πρέπει να δούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις νέες μας φιλοδοξίες. Η έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών διαβιβάζει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα θα ήθελα η νεολαία να αποτελέσει και τον μύτο αυτού του οικονομικού έτους. Η νεολαία είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επενδύσεις λοιπόν για τους νέους σημαίνει επενδύουμε στο παρόν αλλά επενδύουμε και στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για όλους μας σε αυτή τη φάση κρίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο το πέρασμα από, τον ακαδημαϊκό βίο στον εργασιακό βίο. Το 21% των νέων είναι άνεργο. η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει με παθητικότητα το θέμα. Πρέπει να διευκολύνει αυτή τη, τη δύσκολη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο στον ε, ε, κόσμο της εργασίας υπάρχουν επίσης πολύ σημαντικές αλλαγές από τεχνολογικής και δημογραφικής πλευράς. Θα πρέπει λοιπόν η κοινωνία μας να βασίζεται στη γνώση, θα πρέπει να μπορούν να επανακαταρτίζονται, να βρίσκονται σε συνεχή κατάρτιση οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι. Θα έπρεπε λοιπόν η υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης να συγκεντρωθεί στα προγράμματα ακαδημαϊκού τύπου, σε προγράμματα κατάρτισης και θα πρέπει να αυξηθεί η ροή της ανταλλαγής της γνώσης και να έχουμε και εγκυμένη μια πραγματική κινητικότητα. Η κινητικότητα είναι κάτι το θεμελιώδες, είναι μια αξία που την εγγυώνται οι συνθήκες και αποτελεί την καλή βάση για την εσωτερική αγορά. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα στα αγγλικά, γιατί αναπληρώνω και την κυρία Τρίπελ Οπότε έχω έναν διπλό ρόλο. Δεν εξετάζω τώρα μόνο τον προπολογισμό της Κομισιόν, αλλά και των υπόλοιπων ε, θεσμικών οργάνων. Ε, σε αυτή τη φάση της ε, διαδικασίας στόχος μας είναι να σχηματίσουμε μια γενική εικόνα, ειδικά βεβαίως του πλαισίου του προπολογισμού και να δώσουμε κάποιες οδηγίες για τον διοικητικό προπολογισμό διαφορετικών θεσμικών οργάνων και του Κοινοβουλίου πλην Τη Κομισιόν για την οποία βεβαίω μόλι μίλησα. γενικό πλαίσιο. Οι συνθήκε υπό τις οποίες θα υιοθετηθεί ο προϋπολογισμός 2011 είναι πάρα πολύ δύσκολε γιατί βεβαίω το όριο του τίτλου 5 είναι πάρα πολύ περιορισμένο και επειδή η επιτυχής εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας είναι η βασική προτεραιότητα όλων των θεσμικών οργάνων. Η θέση ενισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα αλλάζει την διαδικασία υιοθέτηση του προπολογισμού, γι' αυτό απαιτεί ακόμη στενότερη συνεργασία και διάλογο μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων. Η θεσμική συνεργασία έχει πάρα πολλές επιτυχίες όπως π.χ. οι προσλήψεις, η μετάφραση, και βεβαίως ε, αυτό σημαίνει πως ε, θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματικότητα σε τομείς που δεν είχαμε σκεφτεί μέχρι στιγμής όπως το ΕΜΑΣ, η τηλεεργασία και οι πολιτικές μη διάκρισης. Οπότε το να έχουμε μια στρατηγική μακροπρόθεσμη αποτελεί στόχο και του Κοινοβουλίου και των λοιπόν θεσμικών οργάνων. Οι αβεβαιότητες όσον αφορά το μέγεθος του προϋπολογισμού και τη μορφή του προϋπολογισμού για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και οι αποφάσεις του δικαστηρίου καθιστούν τον τίτλο 5 ακόμη πιο απρόβλεπτο. Συγκεκριμένα για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου οι κατευθυντήριες γραμμές προεδρίου Προεδρείου περιέχουν τα εξής. Πρώτα απ' όλα ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τη δυνατότητα έρευνας των μελών, ε, βιβλιοθήκη, και προσαρμογή των θεσμικών πτυχών ε, στην, της συνθήκη Λισαβόνας. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια νομοθετική αριστεία που είναι κορυφαία προτεραιότητα. Σα ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Uh, Καλωσορίζουμε τον Γιάννους Λεβαντόσκι με τη νέα ιδιότητά του. Πρόεδρε Ερετοί εκπρόσωποι του λαού αρμόδιοι για τα θέματα προϋπολογισμού. Σας άκουσα να ε, εκθέτετε τις ε, ε, προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και σας θυμίζω τις κατευθυντήριες γραμμές που ενέκρινε στις 16 Μαρτίου το Συμβούλιο και έχω να πω ότι συμφωνώ για τα βασικά σημεία. Δεν είναι όμως η συνήθις διαδικασία για δύο λόγους. Ε, που ανέφερε η συγγήτρια του Κοινοβουλίου. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι. Πρώτον, προσαρμοζόμαστε στο νέο περιβάλλον μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εν μέρη έχουμε ήδη προσαρμοστεί, αλλά υπολείπεται έργο γιατί χρειάζεται ε, περισσότερο από ποτέ αγαστή συνεργασία ανάμεσα ε, στα ε, θεσμικά όργανα λόγω της ενίας, μίας ανάγνωσης προβλέπεται για το Κοινοβούλιο, για τον προϋπολογισμό και θυμηθείτε τι έγινε στη συνδιαλλαγή του Οκτώβρη. ελπίζουμε ότι με το νέο χρονοδιάγραμμα θα ε, μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας σε βάση της Διοργανικής Συμφωνίας του 75 και είναι ε, ζωτικός ο ρόλος ε, της ε, συνδιαλλαγής λόγω της μοναδικής ανάγνωσης που προβλέπεται από το Κοινοβούλιο. Αύριο στον τριμερή διάλογο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τους όρους υπό τους οποίους θα διεξαχθεί η συζήτηση και πρέπει να συμφωνήσουμε για τους τεχνικούς όρους της συνδιαλλαγής πριν κινηθεί η επίσημη διαδικασία για τον προϋπολογισμό του 2011. Ο δεύτερος λόγος που εξηγεί γιατί δεν ακολουθούμε τη συνήθη διαδικασία είναι ότι ε, αναβιώ ε, ε, Ξεπερνούμε σιγά σιγά την οικονομική κρίση και πολλά ε, κράτη-μέλη αγωνίζονται να ε, υπερβούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα τους, ε, την υπερχρέωση τους. Υπάρχουν μεγαλύτερες προκλήσεις και περισσότερο από ποτέ πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην χρηστή δημοσιοοικονομική διαχείριση και, στον, στην εξορθολογισμένη υλοποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού. τα Θυμήματα του προυπολογισμου ένα άλφα συγκεκριμένα και 4 έχουν ιδιαίτερη σημασία υπό το φως αυτής της ε, καλύτερης συνεργασίας που χρειάζεται γιατί τέσσερις φορές έχουμε αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές ε, εν των ετησίων διαδικασιών κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να ε, αναθεωρήσουμε ίσως ε, την ε, διοργανική συμφωνία και αυτό θα το συζητήσουμε ταυτόχρονα με την ε, υποβολή του σχεδίου του επόμενου προϋπολογισμού τον Απρίλιο δηλαδή. Η συγγήτρια του Κοινοβουλίου, εμείς εξασκούμαστε για να προφέρουμε σωστά το όνομα της συγγήτριας του Κοινοβουλίου της κυρίας Ζερντεύσκοβγα, μας μίλησε για την έκθεση για τις ε, προτεραιότητες. Ε, σαφέστατα αποδίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στο τμήμα 3 τώρα για την, τα θέματα παιδείας ε, ε, τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την αγορά εργασίας. αυτό είναι αιτιολογημένο γιατί αυξάνεται το αριθμό των ανέργων στην Ένωση. Αλλά εξίσου σημαντικό είναι να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις του σχεδίου ανάκαμψης της οικονομίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες της Ένωσης. Είναι σημαντική η υλοποίηση, αλλά θα επιστρέψουμε η διαδικασία μέχρι το 2011, αλλά εξίσου σημαντική είναι η αποτελεσματική διαχείριση και από αυτή την πλευρά πρέπει να τονίσω ότι φέτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά την προσαρμογή στι συνθήκε τη Λισαβόνα, δεν θα ζητήσει νέε θέσει στον προπολογισμό. Ε, στο κολέγιο των Επιτρόπων θα εγκρίνουμε το σχέδιο στις 27 Απριλίου και όσοι ήθιστε την ίδια μέρα θα ε, υποβάλουμε το σχέδιο ε, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα αρχίσει η διαδικασία για το 2011. Υποσχόμεθα καλή συνεργασία που χρειαζόμαστε γιατί θα έχουμε νέες διαδικασίες και θα τις δοκιμάσουμε για πρώτη φορά φέτος. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Ο κύριος Μπέρμαν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Λεβαντόφσκι, κύριε Πρόεδρε, αναπόφευκτα και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός υφίσταται πίεση. Και στις Βρυξέλλες πρέπει να μετρήσουμε το κάθε ευρώ τρεις φορές πριν το ξοδέψουμε. Κι όμως πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα η αναπτυξιακή βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι στι στοχές χώρε δεν έχουν άλλε ευκαιρίε. Κι όμως η δική του ανάπτυξη θα βοηθήσει τη δική μας κρίση. Η ανάπτυξη δημιουργεί μια αγορά. Μια αγορά που θα αναπτυχθεί γρήγορα. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρώπη αυτά τα χρήματα έξυπνα. Με δάνεια, με μικροχρηματοδότηση, με στήριξη. Επίσης, αν υπάρχουν αυτές οι οικονομικές υπηρεσίες, μπορούν οι άνθρωποι εκεί να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους και ο κύριος Πίμπαλξ, ο Επίτροπος Ανάπτυξης, πρέπει να είναι υπεύθυνο για τον προϋπολογισμό του. Όχι η κυρία Άστον, όπως από είναι το σχέδιο αυτή τη στιγμή. Οι δε επιλογές καταπολέμησης στόχιας δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο των διπλωματικών μας παιχνιδιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Φερνάντες τώρα, πρώτος ομιλητής ξενόματος των ομάδων για δύο λεπτά. Πρόεδρε, αγαπητέ επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα ε, να δηλώσω ικανοποιημένο διότι αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη νέα διαδικασία προπολογισμού το 2011 και αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη νεολαία. Έχει ε, σημασία για το πρόγραμμα Έρασμος για την πρώτη θέση απασχόλησης. Έτσι, ενισχύουμε και την καινοτομία ε, και έχουμε και την ε, ψηφιακή πρόταση. Όλα αυτά συμβάλλουν στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου θα ήθελα να πω ότι το ΕΛΚ ε, τάσεται υπέρ ενός αυστηρού και βιώσιμου προϋπολογισμού ε, όπου θα αιτιολογείται κάθε μία δαπάνη και προτείνουμε λοιπόν να εγκαταλείψουμε ε, το προηγούμενο μοντέλο που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση του προπολογισμού θέλουμε μηδενική βάση, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και εξοικονόμηση πόρων για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα, ε, την πειθαρχία και την αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό και είναι επίγον να έχουμε συγκεκριμένη μακροπρόθεσμη πολιτική ε, για την ακίνητη περιουσία. Θα πρέπει να γνωρίσουμε επίση ε, ποιο θα είναι το ύψο των σταθερών δαπανών να ανάλυση κόστους ωφέλους ε, κάθε μίας πολιτικής ε, που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τονίζουμε ότι η προτεραιότητα του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να είναι η αριστεία ως προς τις νέες νομοθετικές ε, προτάσεις και επίσης θα πρέπει να έχουμε τους απαιτούμενους δημοσιονομικούς πόρους για αυτές τις πολιτικές. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπεται μία μονανάγνωση του προϋπολογισμού και έτσι χρειάζεται καλύτερη συνεργασία, ενισχυμένο σε διάλογος και από πλευράς μας ε, ε, θα δείξουμε ιδιαίτερη αφοσίωση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπαλτσάνη, δυόμιση λεπτά. Η κυρία Μπαλτσάνη, οι κατευθυντήριε γραμμέ για τον προπολογισμό 2011 είναι το πρώτο βήμα για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ένα πολύ συγκεκριμένο βήμα. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμών καταβάλαμε σημαντικές προσπάθειες για να ορίσουμε τις ε, προτεραιότητες προτεραιότητες ισχυρές αναγνωρίσιμες που να δώσουν ορατότητα στην ευρωπαϊκή ένωση με πρώτο στόχος η νέοι η έρευνα η ανάπτυξη όχι μόνο όμως γι' αυτό γιατί ξεκινάμε και για την άσκηση ενορατικών ε, κοινωνικών πολιτικών που θα μπορέσουν να οδηγήσουν στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην αλλαγή του, να σταματήσουν την αλλαγή του κλίματος, να δώσουν δηλαδή μια νέα προοπτική για το μέλλον και να έχουμε πρικοδοτήσεις, κατάλληλες πρικοδοτήσεις χωρίς συμβιβασμούς και χωρίς περικοπές. Είναι ένα πρώτο ρεαλιστικό βήμα αυτό. Το περιθώριο δηλαδή των δημοσιονομικών προπτικών είναι ιδιαίτερα περιορισμένο. Δεν υπάρχουν επαρκή σπόροι, επαρκή κονδύλια για να κάνουμε αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, νέες δράσεις. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό στον τίτλο 1, δηλαδή της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, απασχόλησης. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό θέμα. Ο προϋπολογισμός χρειάζεται και μία ευκαμψία. Θα πρέπει να μπορεί να απαντά έγκαιρα στις απαιτήσεις των πολιτών, στις ανάγκες τους που αλλάζουν. Χρειάζονται λοιπόν προτεραιότητες αλλά και απαράβατοι όροι ούτως ώστε ο προπολογισμό να αποτελεί ένα χρήσιμο μέσο για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Κατάλληλοι πόροι, σίγουρες η υλοποίηση των μελλοντικών στρατηγικών, στρατηγική του 2020 και μία οριστική λύση για ένα μέσο ευελιξίας το οποίο είναι μοναδικό και το οποίο μπορεί να μας επιτρέψει να απαντήσουμε στις μελλοντικές προκλήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκοντμάνης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, Συναδελφοί. Θέλω να τονίσω τρία σημεία. Πρώτον, τα διαρθρωτικά ταμεία, 35% περίπου του προϋπολογισμού, δεν έχουμε τόσο καλές επιδόσεις όσο για την περίοδο 2000 2006. Είμαστε στο 14% σε ποσοστό απορρόφησης. Έχει μειωθεί αυτό το ποσοστό, οπότε αναρωτιόμαστε πώς ε, θα λάβουμε υπόψη, πώς ε, ε, θα υλοποιήσουμε αυτό το κομμάτι του προϋπολογισμού. Αλλιώς δεν θα προφηθούν τα κονδύλια ε, και ε, μπορεί να θα χρειαστεί να μπουν σε αποθεματικό. Επίσης, θα πρέπει να ανακτηθούν ποσά από την προηγούμενη περίοδο 5 δις έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποια κράτη όμως ε, που δεν έχουν ζητήσει την ανάκτηση ε, δεν νομίζω να ζητήσουν ολόκληρο το ποσό και αναρωτιόμαστε θα χρησιμοποιηθούν τελικά αυτά τα κονδύλια ή όχι. Επίσης ε, υπάρχουν δύο πάρα πολύ σοβαρά πράγματα για τις πιστώσεις μεταφορών που μεταφέρονται από ένα χρόνο στον άλλον. το 2009 οι πληρωμές παραδείγματος χάρη ήταν λιγότερες από το 2008 κατά δύο δι και τώρα χρησιμοποιούνται τα κονδύλια, επειδή βασιζόμαστε στις πληρωμές, ε, τοποθετούν λοιπόν σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Δείτε το τμήμα 1α, ε, ό,τι προβλέπετε δηλαδή για την έρευνα. Οι πληρωμές για το 2009 ήταν ε, κατά πολύ χαμηλότερες σε σχέση με αυτές του 2008. Οπότε τελικά ε, θα είναι αρκετά ικανοποιητικά τα αποτελέσματα για να σχεδιάσουμε σωστά τον ε, προϋπολογισμό ε, δεδομένου και των αυξημένων αναγκών. Υπάρχουν αποθεματικά ναι ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Το σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού 2011 μία, περιέχει μία παράγραφο που λέει ότι η χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων δεν θα πρέπει να επιβαρύνει το μη της πολιτικής συνοχής, της διαρθρωτικής πολιτικής ή της γεωργικής πολιτικής. Αυτή είναι μία παρατήρηση η οποία είναι απαραίτητη αν λάβουμε υπόψη μας τους ορισμούς των τίτλων του προϋπολογισμού. Η κρίση πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία λύση θα ήταν η ανανέωση, η καινοτομία. Όμως οι πιο φτωχές περιφέρειες της Ένωσης δεν έχουν τα μέσα για αυτή την καινοτομία, για αυτή την ανανέωση. Άμα θέλουμε λοιπόν εμείς ίσες ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ποντάρουμε στις διαθροτικές πολιτικές και στις πολιτικές συνοχής. Χρειάζεται αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην έχουμε διαφορές μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Ο κύριος Ζιόμπρο. Ο κύριο Πόρτα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρώτα ξεκινάμε τη συζήτηση σήμερα για τι μεγάλε κατευθυντήριε γραμμέ για τον προπολογισμό του 2011 και η προτινόμενη προτεραιότητα είναι η νεολαία. Ε, ε, σε μια περίοδο όπου ε, γίνεται η μετάβαση ανάμεσα στη φοιτησή, στα πανεπιστήμια και την αγορά εργασίας προτείνεται η δημιουργία ενός ε, προγράμματος Εράσμους πρώτη θέση απασχόλησης ε, και το πολιτικό ε, ζήτημα είναι ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες όπως λέμε. Όταν μιλάμε για το Εράσμους πρώτη θέση απασχόλησης τελικά πώς θα υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο με τα κονδύλια του Εράσμους που ήταν για τους φοιτητές ή θα δημιουργήσουμε νέο πρόγραμμα με φρέσκα λεφτά αυτό δεν είναι λεπτομέρεια και δεν είναι λεπτομέρεια να μάθουμε το έρασμό θα είναι για επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, προσωρινές θέσεις απασχόλησης ή για αξιοπρέπειες θέσεις απασχόλησης, ε, για να γίνει σωστή επένδυση, μακροπρόθεσμη επένδυση για τους νέους. Είναι πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας ε, για τους ε, νέους όπως θα έπρεπε να ήταν ή τελικά θα είναι ένα πρόγραμμα για να κρύψουμε την ανεργία. Ε, και τώρα μπαίνουμε στην ε, ε, καρδιά της συζήτησης. Ο προϋπολογισμός το 2011 σημαίνει ότι θα παραμείνει η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να επομιστούμε τις ευθύνες μας. Θα, να χρησιμοποιήσουμε τον προϋπολογισμό το 2011 με σωστό τρόπο, αλλά ο προϋπολογισμός είναι όμοιρος ενός δημοσιονομικού πλαισίου που ισχύει για 7 χρόνια και δεν έχει αναθεωρηθεί παρά την οικονομική κρίση απαιτείται αναθεώρηση του δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλιώ ο προπολογισμό που θα εγκρίνουμε στα τέλη του έτου ε, καταδικάζεται στη μετριότητα του παρελθόντο ακόμη και αν εγκρίνουμε τι βέλτιστε προτεραιότητε που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο ε, και ε, Χρειαζόμαστε λοιπόν ριζική αναθεώρηση και όχι περιθεωρική αναθεώρηση της δομής του προϋπολογισμού. Ευχαριστούμε η κυρία Σεν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, το, η αύξηση κατά 6,5% που προτείνεται στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου το 2011 είναι ακόμη μία ένδειξη του πόσο έχουμε απομακρυνθεί από τον πραγματικό κόσμο και τα συμφέροντα των ψηφοφόρων μας. Πώς θα εξηγήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους αυτά τα πράγματα σε κανονικό καιρό, πόσο μάλλον σε καιρό κρίσης το ότι το κόστος του κάθε ευρωβουλευτή υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια λίρες το χρόνο. Πώς να τους εξηγήσουμε πως θέμε ένα επίπεδο υψηλό και αυτό είναι ο λογαριασμός. Πώς θα το εξηγήσουμε σε αυτούς που χάνουν τη δουλειά τους, ότι εμείς οι ευρωβουλευτές χρειαζόμαστε περισσότερους υπαλληλούς λόγω της συνθήκης Λισαβόνας. Διότι όσοι έχουν εδώ πέρα αξιώματα ε, χρειάζονται περαιτέρω επιδόματα το 15% ανέργων της νεολαίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ή το 45% της νεολαίας που είναι άνεργοι στην Ισπανία δεν αντιλαμβάνονται πώς θα τους βοηθήσει αυτή η αύξηση να βρουν δουλειά. Πολλοί από αυτούς είναι εκπαιδευμένοι και δεν έχουν απλά ευκαιρίες να βρουν δουλειά. Ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να τους απαντήσω. Μπορεί κάποιο να εξηγήσει στους ψηφοφόρους μου πώς το ότι έχουμε δύο έδρες, μία εδώ και μία στο Ρασβούργο, θα τους βοηθήσει να πληρώσουν το στεγαστικό τους και τα, να ταΐσουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι το κόστος των 2 εκατομμυρίων κατά βουλευτή που ανέφερα. Όσον δε αφορά την Κομισιόν, ωραία είναι αυτά που λέμε για επένδυση στην νεολαία, την εκπαίδευση, τις γλώσσες και την καινοτομία για την οικονομική ανάπτυξη κτλ αλλά η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου δεν είναι πολύ παρηγόρη για το πώς ξοδεύονται τα χρήματα αυτά και για το πώς προγραμματίζουμε. Κυρία, κυρία Ανδρέασεν, έχετε ξεπεράσει, έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας. Έχετε το ξεπεράσει το χρόνο σας κατά μισό λεπτό ήδη. Σας ευχαριστώ. Βέρθμαν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι προτεραιότητες του προπολογισμού 2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπό τον αστερισμό της οικονομικής κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση η οποία θα είναι κοινωνικά δίκαιη. Θα επικεντρωθώ σε δύο πράγματα. Ένα μικρό κομμάτι του προπολογισμού αφιερώνεται στην νεολαία εδώ πέρα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο η επένδυση στην νεολαία και κλειδί για την Ευρώπη, γιατί έτσι σκεφτόμαστε την Ευρώπη του αύριο. Και δεύτερον, η υπάρχουσα κατάσταση μας δείχνει ξεκάθαρα το πώς μπορούν να καταστραφούν θέσεις εργασίας. Στρατηγική 2020 έχει έμφαση και στην καινοτομία και έτσι υπάρχουν κάποιες δικαιολογημένες ελπίδες για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να μειωθεί το κοινωνικό χάσμα. Σας ευχαριστώ. Σούριαν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε ότι ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται βαθιές μεταρρυθμίσεις. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι στο πλαίσιο των ετησίων προπολογισμών αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ποιο είναι το πρόβλημά μας. Πρόβλημα ένα, έχουμε λίγη ευελιξία στον προϋπολογισμό μας. Δεν μπορούμε εμείς να αντιδράσουμε στις τωρινές προκλήσεις. Έχουμε λίγο περιθώριο χειρισμών, ελάχιστες δυνατότητες. Η συγγήτρια πρόθεσε μία πρόταση πολύ σημαντική, ε, ισορροπημένη συγγνώμη και διαπίστωσε ορισμένους, ορισμένες προτεραιότητες. Εμείς ελπίζουμε να υποστηρίξουμε το κείμενο το οποίο προτείνεται. Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι ατενίζουμε με ιδιαίτερη προσοχή την νεολαία διότι ε, η νεολαία διατρέχει τον κίνδυνο να απομακρυνθεί από τα ευρωπαϊκά ιδανικά και την Ευρώπη. Η πολιτική συνοχή τώρα, η πολιτική συνοχή ε, δεν είναι φιλανθρωπία. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των ε, ανεπτυγμένων ε, και των ε, υπανάπτυκτων περιοχών της Ένωσης. Πρέπει να μειώσουμε αυτές τις διαφορές. Όταν μία περιφέρεια αναπτύσσεται, αυξάνεται η ανταγωνιστικότητά της και αυξάνεται και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Τα κράτη λοιπόν θα πρέπει να ξοδεύουν τα χρήματα που έχουν στη διάθεσή τους και να ξοδεύονται με αποτελεσματικό τρόπο, με απτά αποτελέσματα, γιατί αλλιώς μόνο σπατάλη θα έχουμε. Να και δύο έδρες του Κοινοβουλίου είναι ένα τεράστιο έξοδο και δεν δίνουν κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Θέλουμε εμείς να μπορέσουμε να, τα χρήματά μας να τα ξοδεύουμε σωστά και καρποφόρο. κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίζω αυτή την έκθεση για τον προ... τις κατευθύνες γραμμές του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό και καλωσορίζω και τη συζήτηση για τις προτεραιότητες μας ούτως ώστε ε, να κάνει σωστά τη δουλειά του το Κοινοβούλιο. Η αρχική έκθεση ήταν ασαφής όπως περιμέναμε, Η γενικόλογη. Βέβαια, ε, οι τροπολογίες, ε, με τις τροπολογίες της Επιτροπής καταλάβαμε ποια είναι τα σημαντικά σημεία. Προσπαθούμε να επιτύχουμε ισορροπία ανάμεσα στις νέες ανάγκες μετά τη Λισαβόνα και την πάγει ανάγκη να κρατήσουμε σε χαμηλό επίπεδο ε, τις δαπάνες ε, γιατί είναι πολύ στενά τα περιθώρια των δημοσίων οικονομικών και θα συμφωνήσουν όλοι ε, πιστεύω. Έχουν κέρια σημασία αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές και δεν μιλάμε μόνο για, την, για τις δαπάνες αλλά και για την εξοικονόμηση πόρων και για τη βέλτιστη χρήση αυτών. Άρα χρειάζεται ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης. Αυτή είναι μια γενικώ αποδεκτή ιδέα και χρειαζόμαστε σωστή πηγή πληροφόρηση για τα κράτη-μέλη ε, και για του πολίτε. Ε, και μέσα από την, ε, τον τηλεοπτικό σταθμό του Κοινοβουλίου οι πολίτε μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία. Επίση, το συνολικό κόστο του προσωπικού, τα, οι δαπάνε για την στέγαση και άλλε τέτοιε διοικητικέ δαπάνε θα πρέπει να εξεταστούν σοβαρά και νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα ε, τη Ένωση. Ε, σχετικά με το κατόφλι του 20% τρόπο συμφωνήσαμε πριν από τόσα χρόνια. Κοιτάξτε, η Επιτροπή Ελέγχου των προπολογισμών ε, πιστεύει ότι θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα ανάμεσα στο Προεδρείο και την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών, αν είναι να αναθεωρηθεί αυτό το ποσοστό και επίση χρειάζεται και διαθεσμικό διάλογο. Δεν πρέπει να γίνει πολιτικό το ζήτημα. Αύριο θα γίνει η ψηφοφορία και ελπίζουμε να βελτιωθούν έτσι περαιτέρω οι κατευθυντήριες γραμμές ε, ούτως ώστε όλες οι διοικητικέ δαπάνες να ενσωματωθούν στο τμήμα 5. Επίσης, ε, οι σε γραμμέ και οι εκτιμήσεις ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν σωστά για να λαμβάνονται και εγκαίρω οι αποφάσει και ελπίζω οι συνάδελφοι να εγκρίνουν αύριο τις σχετικές τροπολογίε. Επίσης, μετά από την συμφωνία που επιτευχθεί για τι σε γραμμέ, υπολείπεται η δυσχερή συζήτηση για τι εκτιμήσει που δημοσίευσε η Γενική Γενική Γραμματεία Εσχάτως και μόνο τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε ουσιαστικά για τις προτεραιότητε και θα γίνει ορθή συζήτηση για να έχουμε την ισορροπία και να λειτουργήσει ε, ορθά το Κοινοβούλιο ώστε να μειωθούν ε, όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται οι δαπάνες. Ε, τώρα ο κύριος Σαχάγκριν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, είναι χαλεπή η οικονομική ε, καιρή ε, και οι κατευθυντήριες γραμμές για το 2011 δεσμεύουν φυσικά και το προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Ως προς το τμήμα 5 και το ποσοστό του 20% έχουμε να πούμε ότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας ορισμένες φορές μπορεί να επιθυμούν αυξημένους πόρους ε, κάποιοι ε, και αυτό ίσως είναι αιτιολογημένο γιατί θα έχει περισσότερες αρμοδιότητες ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 2010 ήδη είχαμε περισσότερους πόρους μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας είναι μηχάνημα αυτόματης ανάληψης για το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σώμα μας να κάνουμε εξοικονόμηση πόρων και να κοστολογήσουμε σωστά τις νέες επιπρόσθετες ανάγκες που έχουμε. Ε, και ακούγονται όλο και περισσότερες φωνές για την αύξηση των επιστώσεων που χρειάζονται οι βουλευτές ε, για να επιτελέσουν τις εργασίες τους. Ε, σωστή ιδέα, αλλά θα έπρεπε να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να ζητάμε συνεχώς περισσότερους πόρους, κυρίως σε αυτή τη δινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει όλες οι χώρες. Πρέπει με επικριτικό πνεύμα να εξετάσουμε τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, είναι δύσκολη η καιρή οικονομικά. Όλοι πρέπει να σφίξουν τη ζώνη και να κάνουν οικονομία. Επιπλέον δεν εμπιστεύονται και πάρα πολύ την ευρωπαϊκή πολιτική οι ευρωπαίοι πολίτες. Έχω λοιπόν δύο προτάσεις για τον προϋπολογισμό. Πρώτα απ' όλα όλοι μας οι ευρωβουλευτές πρέπει για τα 42.000 ευρώ που παίρνουμε για τα γενικά μας έξοδα κάθε μήνα να δώσουμε τον ίδιο λογαριασμό όπως και για τα υπόλοιπα έξοδά μας, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Και νομίζω μαζί με τον συνάδελφο κύριο Στάς θα καταθέσουμε σχετική τροπολογία. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, οι προϋπολογισμοί των εθνικών γραφείων πληροφόρησης του Κοινοβουλίου είναι πολύ περίεργοι αν δούμε το τι γίνεται νομίζω θα μπορέσουν να μειωθούν κατά το 1 τρίτο σε μία περίοδο τριών ετών. Οπότε να είμαστε πιο διάφανοι και να μην εξαιρούμε τους εαυτούς μας. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μπέλντερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο προϋπολογισμός του 2011 μας ε, θέτει ενώπιον των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να αντιληφθούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει χρήματα από τα κράτη-μέλη και έχουμε δύσκολους καιρούς ε, μπροστά μας. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε και οικονομία και καλύτερη χρήση των μέσων. Τώρα, για τις προτεραιότητες που ε, αναφέρει εδώ πέρα ο εισηγητής, ε, κοινωνικά κτλ. Όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Αλλά μιλάτε εδώ πέρα για τη μετάβαση των νέων στην εργασία. Θέλω εδώ πέρα να προσέξετε κύριε εισηγητά, κυρία εισηγητά με συγχωρείτε, τους έθραυστους νέους, τους, την ευαίσθητη νεολαία θα πρέπει να υπάρξει μια ιδιαίτερη φροντίδα τον προηγούμενο μήνα Στη Βουλγαρία είδαμε ένα παράδειγμα το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ θετικό όσον αφορά την ευρωπαϊκή στήριξη στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γκρίφιν για ένα λεπτό. Η πιο σημαντική προτεραιότητα οποιοδήποτε προπολογισμού θα πρέπει να είναι να ξοδεύει κανείς τα λεφτά που έχει. Το να ξοδεύει τα λεφτά αλλού είναι κλοπή. Εν τω μεταξύ γδέρνονται οι Βρετανοί φορολογούμενοι, πληρώνουν 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην Ένωση και ακόμα δεν έχουμε δημοψήφισμα. Εδώ πέρα υπάρχει κάποιο θύμα. 50.000 συνταξιούχοι στη Βρετανία πέθαναν από το κρύο γιατί δεν μπορούσαν να θερμοστούν. Σκοτώνονται οι στρατιώτες μας από τους Ταλιμπάν γιατί δεν έχουν τεθωρακισμένα οχήματα. Χιλιάδες καρκινοπανθείς δεν έχουν να αγοράσουν φάρμακα. 6,4 δισεκατομμύρια λίρες θα κάλυπταν όλες αυτές τις ανάγκες και θα έχτιζαν ακόμα 8 νέα νοσοκομεία και 50 σχολεία. Η προτεραιότητα είναι μία, να σταματήσει το ξόδεμα και να σταματήσουμε να ληστεύουμε την Βρετανία. Για σας είναι προπολογισμό, για τους στρατιώτες, τους καρκινοπαθείς και του συνταξιούχους είναι θέμα ζωής θανάτου. Γκάρι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαιρετίζω τον ε, Επίτροπο Λεβαντόφσκι, παλιό, παλιό φίλο από το Κοινοβούλιο, ο οποίος τώρα έχει αλλάξει έδρανα. Θα ήθελα να μιλήσω για τη στροφή των παραδοσιακών ε, γραμμών του προϋπολογισμού ε, και της παραδοσιακής διαδικασίας. Έτσι μπορεί ο Επίτροπος να ακούσει τις θέσεις του Κοινοβουλίου πριν ξεκινήσουμε στη σύνταξη του πρόχειρου υπολογισμού, του προσχεδίου, του draft budget. Νομίζω ότι αυτά τα οποία λέμε εδώ δεν είναι πια και τόσο διαφορετικά από αυτά που του που του λένε οι γενικές διευθύνσεις και τον πιέζουν από παντού για την υλοποίηση των δικών του στόχων. Εμείς όμως πιέσεις δεν θα σας ασκήσουμε κύριε Λεβαντόφσκι, θέλουμε απλώς να ξέρετε ποιες είναι οι δικές μας προτάσεις. Κάθε μέρα έχουμε νέες προκλήσεις για τον προϋπολογισμό του 2011 έχουμε νέες εντάσεις στην κατηγορία 4 με πολύ στενό περιθώριο που θα ενταθεί γιατί πρέπει να ενισχύσουμε τη στρατηγική της Βαλτικής. Έχουμε προβλήματα. Η Γεωργία όχι μόνο γιατί έχουμε συναπόφαση αλλά γιατί θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε πραγματικά τη συναπόφαση δεν θέλουμε εμείς να φεύγουν χρήματα από, τη Γεωργία για να χρηματοδοτούμε άλλες πολιτικές. Πρέπει επίσης να λύσουμε και το δύσκολο πρόβλημα της κατηγορίας 5 διοικητικά έξοδα διοικητικέ δαπάνε, και θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να κάνει οικονομίες και στον κοινοτικό προπολογισμό και στο Κοινοβούλιο. Αλλά εμείς εκείνο το οποίο είμαστε σίγουρο ότι δεν θέλουμε να κάνουμε είναι να ανεχθούμε τη δημαγωγία αυτών που με τέτοιες πολιτικές πιστεύουν ότι κάνουν πολιτική. Ευχαριστώ. Ο κύριο Φέρμα, αγαπητοί συνάδελφοι και πρώην συνάδελφοι, κύριε Λεβαντόφσκι, καλώ ορίσατε και πάλι. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο και για τι δύο τις εκθέσει. Ευχαριστώ την κυρία Ζερτζεβιέσκα. Ε, ήταν εξαιρετική η έκθεσή τη. Υπάρχουν δύο σημεία για τα οποία οι σοσιαλιστέ υπέβαλαν τροπολογίε γιατί κρίνουμε ότι είναι σημαντικό. Πρώτον, πρέπει να είμαστε σαφείς σχετικά με το ότι οι κλιματικέ αλλαγέ εξακολουθούν να συνιστούν ε, βασική προτεραιότητα. Δεν πρέπει να να, ε, επειδή αποτύχαμε στην Κοπενχάγη, να μην ασκούμε πλέον πίεση για τι κλιματικέ αλλαγέ. Είναι δικό μα καθήκον να βρούμε λύση για το θέμα τη χρηματοδότηση. Δεύτερον, ε, για την στρατηγική Ευρώπη 2020. Απαιτεί η στρατηγική μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει ούτως ώστε να εφαρμοστεί καλύτερα, να υλοποιηθεί καλύτερα η στρατηγική. Πρέπει να είμαστε επιθετικοί για να αναπτυχθεί η οικονομία μας και να προστατεύσουμε και την κοινωνική διάσταση της πολιτικής. Ε, σε αυτό το τομέα χρειάζεται περισσότερη ουσία ε, χρειάζονται μεταξύ άλλων πρώτον σαφές μήνυμα προς τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο ότι δηλαδή θα είναι απαραίτητο να αναθεωρήσουμε το κατόφλιο του προϋπολογισμού για τα επόμενα τρία χρόνια κυρίως στο τμήμα 1 του προϋπολογισμού δηλαδή για την ανάπτυξη για τις θέσεις απασχόλησης για τον προϋπολογισμό του ίδιου του Κοινοβουλίου θα ήθελα να πω ότι πρέπει ε, παρότι έχουμε υψηλέ ανάγκες να λάβουμε υπόψη τους γαλλικούς οικονομικούς καιρούς ε, που βιώνουμε και να αυτοπεριοριστούμε Πρέπει να ενισχύσουμε βέβαια το Κοινοβούλιο και θα ήθελα να τονίσω ε, ότι οι πολιτικέ ομάδε ε, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να σταθούν στο ύψο ε, τη συνθήκη τη Λισαβόνα, να εξοικονομήσουμε πόρου, να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μα κυρίως ε, για το τμήμα 5, για τη διοίκηση, τις διοικητικές δαπάνες. Ε, υπάρχουν μεγάλοι περιορισμοί και συζητούμε τώρα την νέα υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Σίγουρα θα χρειαστούν περισσότερα κονδύλα και υπάρχουν βασικές δαπάνες στο Κοινοβουλίου για, για τις οποίες πρέπει να επιδείξουμε μεγάλο αυτοπεριορισμό. Ευχαριστούμε κύριο Βανόρτη ένα λεπτό. Uh, Κύριε Πρόεδρε, σε καιρού ε, οικονομικά δύσκολου που υπάρχουν περικοπέ στις δημόσιες δαπάνες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να περιορίσουν τις, τους, τις δαπάνες τους και το Κοινοβούλιο πρώτο. Ανταυτού τι κάνει, αυξήνει το προσωπικό του και το κόστος χωρίς να σκέφτεται να περιοριστεί σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Οι νέες προτεραιότητες θα αντιμετωπίζονταν με μειώσεις αλλού, αλλά όχι εδώ μέσα από ό,τι φαίνεται. Οι ευρωβουλευτές κατηγορούνται, αλλά φαίνεται πως και η γραφειοκρατία φταίει και τα περιτά κτίρια. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να δικαιολογούμε τις 94, 94 εκατομμύρια λίρες που δίνονται κάθε χρόνο για αυτοδιαφήμιση του Κοινοβουλίου. Το Europal TV στο διαδίκτυο, να μιλήσουμε για αυτό το νίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας, ότι χρειαζόμαστε επίσης γραφεία πληροφόρηση σε κάθε κράτος μέλος με 40 εκατομμύρια κόστος το κάθε χρόνο. Όταν βεβαίως υπάρχουν 736 ευρωβουλευτές που πρέπει να κάνουν αυτή τη δουλειά και είναι σκανδαλώδες το ότι δεν ζητήσαμε επιτέλους να σταματήσει το Στρασβουργό μια και καλή για να εξοικονομήσουμε αμέσως αμέσως 200 εκατομμύρια το χρόνο. Σας ευχαριστώ κύριε Σομπερμαέρη, δεν είναι εδώ. Η κυρία Γκρέσλε λοιπόν έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, πρώτα απ' όλα να μιλήσω για τον προπολογισμό της Κομισιόν και να σας πω πως η υπηρεσία εξωτερική δράσης μου είναι ιδιαίτερα αγαπητή Δεν αναφέρεται όμω τον προπολογισμό. Είναι αυτό όμω για μας ένα θέμα κλειδί, το πόσο κοστίζει. Είμαι υπέρ του να ανήκει στην Κομισιόν αυτή η υπηρεσία και βεβαίως θα έχει σοβαρές δημοσιονομικές συνέπειες και πολιετής. Δεν μπορεί λοιπόν να κινηθεί εκτός της Κομισιόν. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό το πιο νομικό καθεστώς θα έχει γιατί βεβαίως από αυτό εξαρτάται άμεσα ο προϋπολογισμός και ενδιαφέρον είναι το να δούμε το τι δεν υπάρχει σε αυτόν τον προϋπολογισμό και ελπίζουμε πως θα μπορέσουν σύντομα να μας δώσουν συγκεκριμένα νούμερα οι επίτροποι για την όλη αυτή η υπόθεση το 2011 στην πλευρά της διοίκησης, εκεί που γίνονται τα μεγαλύτερα έξοδα για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, έχουμε τα μικρότερα περιθώρια. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει για εξοικονομήσεις και έχω μία πρόταση. οι διακοπές των υπαλλήλων να μην γίνονται με να μην υπολογίζονται με βάση το σιδηροδρομικό ταξίδι αλλά με βάση το αεροπορικό ταξίδι και με τον ανάλογο χρόνο. Και θα ήθελα λοιπόν να σας πω πως και εμείς θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιες εργασία Τώρα, δεν θεωρώ όμως σωστό να μιλάμε για τα κτίρια. Θεωρώ λοιπόν να ε, πως θα μπορούμε να σας παρακαλέσω να μην καταργήσετε τις θέσεις οποίες έχουμε για τους βοηθούς μας στις περιφέρειές μας γιατί έχουμε εκλογικές περιφέρειες. Αυτά και σας ευχαριστώ. Έρενχάουζερ, για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ. Χρειαζόμαστε μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα διαφορετικό προπολογισμό. Θεωρώ πω χρειαζόμαστε θάρρο για μεγάλε αποφάσει και όχι να ασχολούμαστε με τι μικρέ τεχνικέ λεπτομέρειε. Τρία πράγματα για τον προπολογισμό. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε διαφάνεια. Π.χ. τα διοικητικά έξοδα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ρεαλιστική απάντηση. Δεύτερον, εξοικονομία. Δεν μπορεί να ξοδεύουμε δισεκατομμύρια χωρίς να δούμε το τι γίνεται με την ποιότητα. Π.χ. εδώ πέρα μπορούν να κλείσουν πάρα πολλέ από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Να δούμε τι θα γίνει με το Στρασβούργο ή όλα αυτά τα βήματα χωρίς ε, αρμοδιότητες, π.χ. η ΟΚΕ, η Επιτροπή των Περιφερειών. Τι κάνουν. Επίσης, να επιστραφούν τα λεφτά εκεί που ανήκουν στου φορολογούμενου. Εννοώ βεβαίω να προωθήσουμε λογικά έργα με αυτό. Να έχουμε π.χ. ένα πραγματικό ερασμό για τους μαθητές. Πρέπει λοιπόν όλοι να βρούμε θάρρο για να τα κάνουμε αυτά. Ευχαριστώ. Σκέρσκι για δύο λεπτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει νέες αρμοδιότητες με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ήρθε η ώρα λοιπόν της συναπόφασης, πρέπει όμως να αρχίσει να λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Θα είναι πολύ σημαντικό ε, σημαντικό το 2011 και επόμενες χρονιές για τον ορισμό της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Μόνο η συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε μία διαδικασία που θα ανταποκρίνεται στις διατάξεις της συνθήκης. Υποστηρίζω την έκκληση για αύξηση του προϋπολογισμού της Ένωσης ε, από τη Λισαβόνα και μετά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκπληρώσει το ρόλο του. Χρειάζεται την ανάλογη πρικοδότηση. Η σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυξάνεται. Χρειάζεται, χρειαζόμαστε και εμείς οι βουλευτές μεγαλύτερη υποστήριξη από εμπειρογνώμονες και όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι επιπληρωμή. Μια άλλη πλευρά της έκθεσης είναι το να έχουμε περισσότερες επενδύσεις για την νεολαία. Χρειάζεται λοιπόν να επενδύσουμε στην παιδεία που αποτελεί και τη βάση της σύγχρονης κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανταγωνιστεί με τις Ηνωμένε Πολιτείε και άλλες ε, μεγάλες ε, δυνάμεις, βιομηχανικές δυνάμεις στο τεχνολογικό τομέα. Πρέπει να επενδύσουμε στην τεχνολογία για να ανακτήσουμε την καθυστέρηση. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την φτώχεια. Πρέπει να ενισχύσουμε το μέσων επισητισμού ε, θα πρέπει να επιβάλλουμε το ποτήρι γάλας ή τα φρούτα και τα λαχανικά στο σχολείο. Μιλάμε πολλά για εκπαίδευση, μιλάμε, ε, λέμε πολλά για την οικονομία, λέμε πολλά για τη γνώση. Σήμερα έχουμε και τη στρατηγική 2020. Έτσι λοιπόν ήδη σε αυτούς τους προσανατολισμούς του προϋπολογισμού πρέπει να ορίσουμε την προϋκοδότηση και τη χρηματοδότηση αυτής της στρατηγικής για να μπορέσει να πετύχει αυτή η στρατηγική χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις σε επίπεδο συνοχής και πρέπει να παλέψουμε για να καταπολεμήσουμε τα τις επιπτώσεις της κρίσης. Λοιπόν, ευχαριστώ την κυρία Γιαζεύκα για τις καινότομες προτάσεις. Καρβαλιό, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η νεολαία, η έρευνα και η καινοτομία είναι στον πυρήνα του νέου προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να επενδύσουμε στη νεολαία και στο μέλλον. Η παιδεία, η επαγγελματική κατάρτιση, η μετάβαση του από το εκπαιδευτικό σύστημα προ την αγορά εργασία. Να οι βασικέ ανησυχίε που εγγράφονται στον προπολογισμό. Ε, και οι νέοι πλήττονται, λένε και περισσότερο, από την ανεργία. Οπότε το πρόγραμμα κινητικότητα, ε, έρασμο, ε, πρώτη θέση απασχόληση είναι μια επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα στο μέλλον. Χρειαζόμαστε με μια σαφή διασύνδεση ανάμεσα ε, στο σύστημα παιδείας ε, και την αγορά εργασίας. Ε, οπότε αυτό το πρόγραμμα Εράσμους, πρώτη θέση απασχόλησης που συνυποβάλαμε τον κύριο Φερνάνδης βασίζεται στις εξής αρχές. Πρώτον, επιπρόσθετη χρηματοδότηση των υφιστάμενων προγραμμάτων στον τομέα της παιδείας, της έρευνας και καινοτομίας. Δεύτερον, κάθε δράση θα έχει μια επιπρόσθετη κατάρτιση και στη συνέχεια θα υπάρχει σύμβαση με καινοτόμα επιχείρηση ε, που θα συγχρηματοδοτείται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ε, ε, μέσα στον προϋπολογισμό επίσης βλέπουμε την καινοτομία, την έρευνα και την ψηφιακή ατζέντα, περαιτέρω προτεραιότητες δηλαδή για τον νέο προϋπολογισμό. Ε, θέλουμε να αναπτυχθούν ε, νέες καθαρές ε, καινοτόμες τεχνολογίες γιατί έτσι θα επιτύχουμε την ανάκαψη της οικονομίας και θα γίνουν πιο δυναμικές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το κλειδί ούτως ώστε η Ευρώπη να ανακτήσει την ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστούμε βάσει της διαδικασίας Catch the Eye τώρα. Ο κύριος Μπόρις, ένα λεπτό. Κύριε Επιτροπέ, Κυρία Ισηγήτρια, θέλω να σας συγχαρώ για αυτή την καταπληκτική έκθεση. Η οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Και η έκθεση απαντάει σε μία ερώτηση. Πώς να εγγυθούμε την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν χρηματοδοτεί την νεολαία που είναι και το πιο μεγαλόπνο σχέδιο για το μέλλον. Για την νεολαία πρέπει να ενισχύσουμε τις ψηφιακές τεχνολογίες ε, για το μέλλον της Ευρώπης, να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως στις μονεκτικές περιοχές. Υπάρχει και κάτι άλλο, η κινητικότητα των επενδύσεων. Παίζει σημαντικό ρόλο, συγγνώμη, οι επενδύσεις για την κινητικότητα. Χρειάζεται χρηματοδότηση των μεγάλων δικτύων. Ευχαριστώ την ε, Επιτροπή λοιπόν που ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Τικάου, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κύριε πίτροπε, ο προϋπολογισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις νέες αρμοδιότητες της Ένωσης οι προτεραιότητες είναι να παραμείνουν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν καινούργιε. Πρέπει να έχουμε μια βιομηχανική πολιτική ευφύ και φιλόδοξη. Δεν μπορούμε εμείς ε, να χρηματοδοτούμε τη βιομηχανία μόνο με το 15% του ΕΠ. Πρέπει λοιπόν να δοθούν στα κράτη-μέλη το 2011 οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις μετά από τη μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών προοπτικών 2000 μέχρι το 2013. Πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, πρέπει να επενδύσουμε στον τομέα της υγείας, πρέπει να επενδύσουμε στις υποδομές των μεταφορών και όλα αυτά πρέπει να τα δούμε στον προϋπολογισμό. Κύριος Φερέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Η οικονομική και η κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί για το 2011 να θεωρήσουμε άρδιν τι προτεραιότητε που είχαμε στου προηγούμενους προπολογισμού και στον τωρινό το 2010. Πρέπει να εξυπηρετούνται συγκεκριμένες πολιτικές ε, και ξέρετε ότι έχουμε πάνω από 23, 23 εκατομμύρια ανέργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πλήττονται από τη φτώχεια εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ε, ε, λόγω του πολιετού δημοσιονομικού ε, πλαισίου και ε, που αντιστοιχεί στο 37% του ΑΕΠ της Ένωσης ε, και πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα, στην παιδεία και στον πολιτισμό και με οι μελλοντικοί προπολογισμοί πρέπει να εξυπηρετούν την οικονομική και κοινωνική συνοχή και να παραμένουν σε οι συνθήκες κενέ περιεχομένου. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το προπολογισμό ως μέσο για να εξυπηρετήσουμε ε, την κοινωνική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή ε, και να μην ε, επιτρέπουμε να διεξάγονται πόλεμοι, να ακολουθείται μερκαντιλιστική πολιτική μέσα από του προπολογισμού που εμεί εγκρίνουμε. Χρειάζεται άρτην αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών του πολιετού δημοσιονομικού πλαίσιου. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Σομπερμάιερ, ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ αναφέρομαι στο 5 για τη στρατηγική για τα κτίρια. Μια στρατηγική επιτυχής δεκτήρια είναι σημαντική. Θα πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον και αποτελεσματική όσον αφορά την χρήση ενέργεια και το κόστος. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον ε, είναι λογικό να έχουμε τρει τόπου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Το τεράστιο κόστο δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε ένα του φορολογούμενου σε μια εποχή οικονομική κρίση. Θα πρέπει να γίνει μια ει ε, ανάλυση του κόστους και να τη διαθέσουμε και στους πολίτες. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συγκεντρωθεί σε ε, μία έδρα και εγώ θα έλεγα ότι το Στρασβούργο θα ήταν η καλύτερη λύση λόγω του ότι οι τη άλλη, οι Βρυξέλλες ε, πνίγονται στην εγκληματικότητα και όπως το παραδέχεται ο κ. Στίλεμανς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2011 θα πρέπει να στηρίξει περισσότερο τις πολιτικές υπέρ της νεολαίας. Πρέπει να στηρίξουμε τους νέους και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω να σας υπενθυμίσω εδώ ότι στη Ρουμανία ένα από τα προγράμματα που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση για να στηρίξει την νεολαία είναι υπέρ 100.000 κατοικιών για τους νέους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Η υποτροφία Έρασμος επίσης κοντεύει τα 3 εκατομμύρια να φτάσει. Όμως πρέπει να χρηματοδοτείται καλύτερα το Έρασμος Μούντους διότι μόνο έτσι περισσότεροι νέοι ερευνητές τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τρίτες ε, χώρες και από τη Μολδαβία θα μπορέσουν να σπουδάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως νέα Ευρωβουλευτής στηρίζω την πρωτοβουλία Εράσμους και θέλω να δώσουμε περισσότερα μέτρα στήριξης υπέρ των νέων. Και ευχαριστώ και την Επιτροπή για τη στήριξή στα ενεργειακά προγράμματα υπέρ της Ρουμανίας. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επίτροποι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση στα κράτη-μέλη και συγχρόνως πρέπει να δώσουμε πολύ προσοχή στον προπολογισμό του 2011. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση και όταν πρόκειται για τη στήριξη υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, γιατί αυτέ προσφέρουν θέσει εργασία στου πολίτε μα. Θέλω λοιπόν να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις αυτές και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες μέσω των οποίων προσφεύγουν σε χρηματοδοτική στήριξη. Δεν πρέπει να βαραίνουμε περισσότερο τη γραφειοκρατία. Αντίθετα, πρέπει να τι βοηθήσουμε γιατί και αυτέ μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει ιδιαίτερα να δώσουμε προσοχή επίση στι μεταφορέ και στα προγράμματα υποδομών, όπω επίση και σε προγράμματα υπέρ τη ενέργεια. Αυτοί οι στόχοι πρέπει να αποτελέσουν την προτεραιότητά μας για τον προπολογισμό του 2011. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας τα οποία με βοηθούν να κατανοήσω καλύτερα τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2011. Αυτό το οποίο φάνηκε ξεκάθαρα ακούγοντάς σας σήμερα το βράδυ. Αυτό λοιπόν που ήταν ξεκάθαρο για μένα ήταν ότι πολλοί ομιλητές υπογραμμίζουν πώς σχεδιάζουμε τον προπολογισμό του 2011 κάτω από έκτακτες συνθήκες μετά την οικονομική κρίση όπου πολλές χώρες αντιμετωπίζουν προκλήσεις δημοσιονομικές ακόμα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πίεση στον προπολογισμό, κάτι το οποίο πιέζει και υπέρ της διαφάνειας του προπολογισμού και χρηστή διαχείριση. Αυτό το είπαν και Βανόρντεν, Μπέργουεν, Χάτλου κλπ. Όμως, όταν δεν έχουμε αρκετού πόρου, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι σωστά να καθορίσουμε τι προτεραιότητε μα. Η αίσθησή μου μετά τη συζήτηση είναι ότι η νεολαία πρέπει να στηρίζεται. Και τη στηρίζουν την νεολαία τόσο οι νέοι όσο και οι λιγότερο νέοι ευρωβουλευτέ του σώματο. Άρα, όντω, είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για τον προπολογισμό του 2011 σύμφωνα με την πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο. Αυτό το οποίο επίση χρειάζεται είναι ποιότητα και καλή εφαρμογή, καλή χρήση των πόρων. Ο κύριο Κόντμαντ, ο κύριο Σούλιαν ε, μιλήσανε για τη συνοχή. Ναι, Ητανε χαμηλού επίπεδου το 2009 και 2010. Θα έπρεπε να επιταχυνθεί το 2011 ως μέτρο κατά της κρίσης, για να βγούμε από την κρίση. Όμως η έρευνα επίσης χρειάζεται ρυθμίσεις καλύτερες που να την στηρίζουν και να την ενισχύουν. Αυτό το οποίο επίσης ήταν ξεκάθαρο για μένα ακούγοντας τη συζήτησή σας ήταν ότι το Κοινοβούλιο αντιλαμβάνεται πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ελιγμών στον προπολογισμό. Κύριο Σονταρίκα, Φέρμου και άλλοι το υπογράμμισαν ε, αυτό. Ότι έχουμε πολύ μικρό περιθώριο ελιγμών. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ελαστικοί στην εφαρμογή του προπολογισμού. Συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ με το συμπέρασμα αυτό. Είναι και Κρέσλε, ως συνήθως έχει δίκιο που λέει ότι οι υπηρεσίε εξωτερική δράση δεν έχουν πρικοδοτηθεί αρκετά. Ναι, αλλά για να δώσουμε χρήματα χρειαζόμαστε ποσά. Και χωρί ποσά, χωρί νούμερα, δεν μπορούμε εύκολα να αποφασίσουμε για τον προπολογισμό. Αλλά αυτό θα γίνει φέτο, εφόσον η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων αρχίσει να λειτουργεί. Οπότε, ε, περιμένω με ανυπομονησία την αυριανή συζήτηση στον τριμερή διάλογο και μετά να ξεκινήσει η πραγματική συζήτηση που θα οδηγήσει και σε καρποφόρα σε διαλλαγή για τα ποσά του 2011. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Να δώσω το λόγο τώρα για να ολοκληρώσει η κυρία Γεντρεζεύσκα. Η κυρία Σετρεζεύσκα, λοιπόν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα όλες τις απόψεις που ακούστηκαν σε αυτή τη συζήτηση και χαίρομαι που συμφωνείτε με τις βασικές προτεραιότητες που έχουμε θέσει για τον προπολογισμό. Να υποστηρίξουμε καταρχάς τους νέους. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που το υποστηρίζετε αυτό και αυτό μου δει κίνητρο να κινηθώ με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, ακόμα μεγαλύτερη. Πολλοί από εσά σωστά είπατε ότι έχουμε ελάχιστα περιθώρια ελιγμών. Γι' αυτό θα ήθελα να επαναλάβω την έκκλησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πραγματοποιήσει την αναθεώρηση, την ενδιάμεση αυτή αναθεώρηση του πολιτούς ε, αυτού δημοσιονομικού πλαισίου. Είμαστε στο πέμπτο χρόνο του πολιτού πλαισίου και έγκυκε η ώρα συναγωγής συμπερασμάτων μετά από τετραετία εμπειριών. Είναι σαφέστατο ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επλήγημεν διαφορετικά στα διάφορα κράτη-μέλη και προσπαθούμε να εξέλθουμε από την κρίση και να αναζωογονήσουμε τις οικονομίες μας. Έχουμε κάποιους πόρους για ανάπτυξη, για έρευνα, για την νεολαία, για την ενιαία αγορά, για τις ελευθερίες και είναι όμως ένα μικρό τμήμα του προπολογισμού τα χρήματα που διατίθενται για όλα αυτά. Αν περικόψουμε τον προπολογισμό, αυτό θα ήταν ο λανθασμένο χώρο από τον οποίο θα πρέπει να γίνουν περικοπέ. Πολλοί από εσά είπατε ότι οι νέοι είναι το μέλλον μας. Αυτό είναι ηλίου φαϊνότερον. Αλλά έχουμε και εδώ νέους εδώ και τώρα που δεν ζουν στο απόμακρο μέλλον, αυτοί οι νέοι ζουν σήμερα στην Ευρώπη. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουν ανάγκες. Θα ήθελα να πω μερικά λόγια επίσης για την ευρύτερη προοπτική για μια γενικότερη προσέγγιση, ευρύτερη προσέγγιση όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όταν αναφερόμαστε στους νέους. Δεν μιλάμε μόνο για άμεση υποστήριξή τους, αλλά είναι και άλλη διάσταση, η διάσταση της παιδείας. Και εδώ είναι σαφέστατη υποστηθέμενη αξία που μπορεί να δοθεί. Να μην λησμονούμε ότι έχουμε μία κοινή Ευρώπη, ενιαία Ευρώπη και ελεύθερη κινητικότητα, ελεύθερη μετακίνηση αφορά όχι μόνο ε, τους ανθρώπους αλλά τις ιδέες και τις σκέψεις. Θα ήθελα να συνοψίσω και τη συζήτηση για τον προπολογισμό που διεξήχθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα υπό την ιδιότητα του συναδέλφου που απουσιάζει σήμερα, που είναι συγγητής, είναι σαφέστατο ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε κάποια μέτρα λιτότητας Πρέπει να γίνουν κάποιες περικοπές, θα πρέπει να δικαιολογηθούν οι δαπάνες μας και αυτή η πειθαρχία, αυτή η λιτότητα, αυτή η αυστηρότητα ισχύει για όλους και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντικατοπτρίζεται στην έκθεση που εκπονήθηκε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών συζητούμε το θέμα αυτό τέτοια ώρα που είναι αργά. Ελπίζουμε να μην τα σπατάλει χρόνο, να μην θεωρήσετε ότι σπαταλήσαμε το χρόνο μας. Ελπίζω να μην είναι ότα κοφά τα ότα του Επιτρόπου. Ε, θα πρέπει να θυμάται ότι κάποτε καθόταν σαν συνάδελφος ανάμεσά μας. Και ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση και οι ιδέες μας θα αντικατοπτριστούν στην πρόταση που πρόκειται να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 του Απριλίου. Θα χαιρόμουν πολύ αν έβλεπα αυτές τις ιδέες στο σχέδιο κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτω ώστε να μην πρέπει να επαναλάβουμε τα υποθέντα σήμερα. Ευχαριστώ. Η κοινή συζήτηση περατώθηκε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, στην επόμενη συζήτηση, θα ήθελα να ακούσω κάποια ανακοίνωση. Προάσπιση ασυλίας ενός βουλευτή.